Chers Αγαπητοί συνάδελφοι. Καλησπέρα. Μάλλον όλοι είναι εδώ. Αγαπητοί συνάδελφοι, καλησπέρα. Καθίστε παρακαλώ. Για τη συνεδρίασή μας αφορά την ψηφοφορία μας, στη συνεδρίαση. Έκθεση της Επιτροπής. Παρακαλώ να καθίσατε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ τις ομάδες που κάνουν τις θέσεις τους. Η συνεδρίαση ίσως να είναι μακράς διαρκείας. Έχουμε πολλά. Ανάλογα με το πώς θα πάει η ψηφοφορία θα δούμε. Ευχαριστώ για την παρουσία σας, πολύ εδώ απόψε. Θέλω να ευχαριστήσω και να συγχαρώ την συνεισηγήτρια, του σκιώδης των διαφόρων ομάδων, τους συντονιστές ε, και τις ομάδες για την προετοιμασία της απόψινής συνεδριάσεως, την ψηφοφορία της εκθέσεως. Πριν πάμε στην ημερήσια διάταξη. Ενός λεπτού σιγή θα παρακαλούσα να τηρήσουμε εις μνήμη των επιθέσεων της 13ης Νοεμβρίου, σαν άμνηση των επιθέσεων της 13ης Νοεμβρίου, στο Μπατακλάν, στο Stade de France και στο τεράστιο που έγιναν εδώ και τρία χρόνια σήμερα, με 137 νεκρούς, 413 τραυματίες και 99 πολύ σοβαρά τραυματίες. Αν έχει την καλοσύνη, ε, ενός λεπτού σιγή παρακαλώ. Je vous remercie. Λοιπόν, έγκριση τη ημερήσια διάταξη ω ήθιστε, αν δεν υπάρχει αντίρρηση, αποχέ θεωρείται συγκεκριμένη ημερήσια διάταξη. Το σημείο 2 τη ημερήσια διάταξη είναι αφιερωμένο στην έγκριση των πρακτικών των διαφόρων συνεδριάσεων τη επίτροπή που έχετε λάβει τα πρακτικά αυτά. Δεν υπάρχει αντίρρηση, κάποια ένσταση εποχή θεωρώ ότι πρόκειται περί εγκεκριμένων τη 4η και 9 ε, Νοεμβρίου του 2018. Είναι τα πρακτικά σημείων 3. Ε, ε, εντάχει, ανακοινώσει Προεδρία πριν περάσουμε στην ημερήσια διάταξη της ψηφοφορία. Είμαστε στο τέλος των εργασιών μας, εντός των προθεσμιών της θητείας. Να πω ότι σε αυτή τη συνεδρίαση απόψε θα έχουμε και διαρμηνία ενεργό και παθητική, γαλλικά, γερμανικά, ιταλικά, ολλανδικά, αγγλικά, ελληνικά, ισπανικά, πορτογαλικά, ουγγρικά, πολωνικά και ρουμανικά. Μπορούμε να έχουμε και διαρμηνία δανέζικη, αλλά μόνο σε παθητική μορφή. Ευχαριστώ τους συναδέλφους για την κατανόησή τους. Ζητώ συγγνώμη στους συναδέλφους που δεν έχουν τη γλώσσα τους στη διερμηνή απόψε. Πάμε στην ψηφοφορία. Αφορά διαπιστώσεις και συστάσεις της ειδική Επιτροπής για την Τρομοκρατία. Σας προτείνω για την καλή ροή της διαδικασίας και για αποτελεσματικότητα της ψηφοφορίας να προχωρήσουμε γρήγορα μέσω ηλεκτρονικής ψηφοφορίας ούτως ώστε να μπορούμε να έχουμε και αποτελέσματα αδιαμφισβήτητα και σαφήνεια στην ψηφοφορία. Καμιά φορά δεν είναι σίγουρα τα πράγματα, λέει η Πρόεδρος, και έτσι μπορούμε να προχωρήσουμε πιο γρήγορα. Αν συμφωνείτε, ας ξεκινήσουμε. Αμέσως. Προήμιο. Ξεκινάμε την ψηφοφορία. Le vote Πέρας ψηφοφορίας. Ο κ. Ντανζάν, δεν είμαι σίγουρος ότι είναι και ο πιο γρήγορος τρόπος αυτός. Θα επιτρέψει, λέει Προέδρος, να υπάρξει μεγάλη σαφήνεια. Και προτείνω αυτό να κάνουμε. Πρώτα απ' όλα να κάνουμε κάποια επαλήθευση ότι δεν έχουμε παραπάνω μέλη από ό,τι πρέπει. Υπάρχει ένα μέλος του ΕΛΚ περισσότερο. Ένα συνάδελφος του ΕΛΚ περισσεύει. Alors, un PPE de trop. C'est bon Είμαστε εντάξει. Η γραμματεία μου λέει ότι πάντα έχουμε ένα μέλος του ΕΛΚ παραπάνω. Όλα εντάξει τώρα. Πολύ ωραία. Ας προχωρήσουμε αν συμφωνείτε λοιπόν. Να ξανακάνουμε τη δοκίμη. Διότι η γραμματεία έχει καταγράψει 31 μέλη, ένα μέλος του ΕΛΚ παραπάνω. Ξαναξεκινάμε. Προήμιο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ένας παραπάνω πάντα, αγαπητοί συνάδελφοι. Εντάξει είμαστε τώρα. Πολύ ωραία. Έτσι φαίνεται ότι είναι όλα εντάξει τώρα. Η οριζόντια τροπολογία άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. ΕΕΦ EF1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική EF2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας αυτής. Εγκρίνεται. 2. Παράγραφος 2α νέα. Τροπολογία 644. Άρχεται η ψηφοφορια περας αυτης εγκρινεται παραγραφος 2 α νεα τροπολογια 644 αρχεται η ψηφοφορια

Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 651 της παράγραφος 3 πάντα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 652 Παράγραφος 3α πάντα, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική IF3, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 654. Ονομαστική ψηφοφορία αυτή 654 και 56 για την παράγραφο 3α νέα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτονται. 660 παράγραφος 4α άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας αυτής εγκρίνεται. 662 για την παράγραφο 4α άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 661 παράγραφος 4α νέα άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 72α νέα, τροπολογία 1199, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Αιτιολογική σκέψη εα νέα, τροπολογία 44, άρχεται η ψηφοφορία. καταπίπτει. Ζητώ συγγνώμη, λέει Πρόεδρος. Τετρα. Καταπίπτει αν οι 662 και 661 δεν εγκρίνονται, οπότε καταπίπτει αυτή. 403 πάμε τώρα. Άρχεται η ψηφοφορία. Καταπίπτει. Πάμε στα 403. Άρχεται η ψηφοφορία για την 403. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική IF4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. εγκρίνεται. Τροπολογία 663. Άρχεται η ψηφοφορία για την παράγραφο 4α νέα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 4α. Τροπολογία 664. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Παράγραφος 4β νέα, τροπολογία 665 και 68, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική ΤΑΦ 1, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Πάμε στην 672, την παράγραφο 5α νέα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 673 και 86 ψηφίζονται ομού για την παράγραφο 5α και τη ολική σκέψη JA. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική ΤΑΦ 2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 684. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Συμβαστική ΤΑΦ 3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. ΤΑΦ 4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 710 για την παράγραφο 9 σε 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Παράγραφος 8 σε 9, τροπολογία 704. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Τροπολογία 705 για την παράγραφο 9α. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Παράγραφος 10α νέα τροπολογία. 706 για την παράγραφο 9α νέα. Για την 706 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. 9β νέα παράγραφος, τροπολογία 708, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 709, για την παράγραφο 9 σε 9, ψηφίζουμε. Τέλος ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Σημαστική ΤΑΦ 5, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Πάμε στην 903 για την παράγραφο 26α. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Παράγραφος 9D, νέα. 711. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 729 για την παράγραφο 10α. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 727 για την παράγραφο 10α. Καταπίπτει. Λοιπόν, ψηφίζουμε την 727. Τέλος. εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στο συμβιβασμό R1, ριζοπαστικοποίηση 1, άρχεται, πέρας, εγκρίνεται. Συμβιβασμός R2, ψηφίζουμε, ελπίζω να μην πηγαίνω πολύ γρήγορα λέει η Πρόεδρος, πέρας της ψηφοφορίας, Πέρας λέω εγκρίνεται συμβιβαστική R3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται συμβιβαστική R4. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται συμβιβαστική R5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 880 επί της παραγράφου 25α νέο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Τροπολογία 881 επί της παραγράφου 25b νέο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική R6 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 770 επί της παραγράφου 14α νέο άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική R7 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική R8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 789 επί της παραγράφου 15b νέο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και απερίφθη η τροπολογία. Συμβιβαστική R9, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική R10, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 814, επί της παραγράφου 17α νέο, Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και απερίφθη η τροπολογία αυτή. Συμβιβαστική R11. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 823 ε, απερίφθη. 8, 16, 17, 18 τροπολογίες ταυτόσιμες άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Ο... 823 Τροπολογία 823, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Τροπολογία 823, απερίφθη. Τροπολογία 822, άρχεται. Πέρας. Απερίφθη. Συμβιβαστική R12, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 830 επί της παραγράφου 19α νέο, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική R13. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική R14. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. Συμβιβαστική R15. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας Εγκρίνεται. Συμβιβαστική R16. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. Τροπολογία 865 και τροπολογία 867 είναι ταυτόσιμες. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. 864 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 866 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Συμβιβαστική R17 άρχεται η ψηφοφορία. πέρας εγκρίνεται. Συμβιβαστική R18, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και εγκρίνεται. Συμβιβαστική R19, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Συμβιβαστική R20, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται τροπολογία R21, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται ε, τροπολογία συμβαστική R22, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται Τρο, συμβαστική R23, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. R24. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. Συμβιβαστική R25. Ας αρχίσουμε να ψηφίζουμε. Ας σταματήσουμε τώρα να ψηφίζουμε. Εγκρίνεται. R26. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 925. Επί της παραγράφου 28α νέο ναι, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Συμβιβαστική R27 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική R28. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική R29. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. Συμβιβαστική R30. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική R31. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. Περνάμε στην τροπολογία 963 επί της παραγράφου 30α νέο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 950, άρχεται η ψηφοφορία. Αντέχετε, ρωτάει η πρόεδρος στη γραμματέα. Καλά πάω, λέει. 951. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Συμβιβαστική R32. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην συμβαστική για την συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών, CIE, συμβαστική 1, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας, εγκρίνεται. CIE 2, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας, εγκρίνεται. Συνεργασία και ανταλλαγή πληροφοριών 3 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 981 επί της παραγράφου 33α νέο άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας απερίφθη. Συμβαστική CIE 4 άρχεται η ψηφοφορία πέρας και εγκρίνεται. CIE CI5 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. CIE CI6 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. CIE CI7 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται. Τροπολογία 1197 επί της παραγράφου 72α νέο άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και απερίφθη. Τροπολογία 1008 επί της παραγράφου 37α νέο άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας απερίφθη. Τροπολογία 1009-1009 επί της παραγράφου 37α νέο άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Απερίφθη. Συμβιβαστική CIE 8 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Τροπολογία 1014 επί της παραγράφου 39 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Συμβιβαστική CIE 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική CIE, CIE 10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και εγκρίνεται. Συμβιβαστική CIE 11, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1023. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και απερίφθη. Τροπολογία 1024, 1025, 1026 ταυτόσημες. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 1029 και 1030 ταυτόσημες. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Ψηφίζουμε τώρα την τροπολογία 1031 επί της παραγράφου 42. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 1032. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1033 επί της παραγράφου 42α νέο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1034-1035, ταυτόσημες, πάντα για την παράγραφο 43, άρχεται, πέρας, απεορρίπτεται. Συμβιβαστική CIE 12, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας, εγκρίνεται. Συμβιβαστική CIE 13, άρχεται η ψηφοφορία, Πέρας εγκρίνεται. Τροπολογία 1049 επί της παραγράφου 45α νέο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και απορρίπτεται. Τροπολογία 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 5056. επί της παραγράφου 46 είναι ταυτόσιμες και απομένως ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1059. 1060, 1061, επί της παραγράφου 47, ταυτόσιμες ψηφίζονται λοιπόν μαζί, άρχεται η ψηφοφορία, Πέρας. Απερίφθη. Συμβιβαστική CIE 14, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 1067, επί της παραγράφου 48α νέο, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Συμβιβαστική CIE 15. CIE 15, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. Τροπολογία 1074, επί της παραγράφου 50. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας απερίφθη. Τροπολογία συμβιβαστική CIE 16 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Τροπολογία 1079 της παραγράφου 52 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας απερίφθη. 1080, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας, απερίφθη. 1081, άρχεται η ψηφοφορία, πέρας, απερίφθη. Η συμβιβαστική ΣΥΕ 17, ε, άρχεται η ψηφοφορία, Πέραση ψηφοφορία εγκρίνεται. Σε 18 ε, άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία εγκρίνεται. Τροπολογία ε, 1095 άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορία εγκρίνεται. Συμβαστική σε 19 ε άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Ε, 1188 ε, άρχεται ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 10 98 άρχεται η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Η συμβαστική σε 20 άρχεται η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται. Σε 21 άρχεται η ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας, εγκρίνεται τροπολογια 11.14 της παραγράφου 56β σε δύο τμήματα. Μα, νομίζω ότι είμαι αρκετά γρήγορη, λέει ο πρόεδρος. Δεν μπορώ να πάω πιο γρήγορα. 1114 επί της παραγράφου 56β πρώτο τμήμα. Πέραση τις ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Δεύτερο τμήμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. Συμβαστική σε ΙΕ 22 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 11.22 επί της παραγράφου 57 β άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβαστική σε 23. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική σε 24. Άρχεται η ψηφοφορία. ψηφοφορία. ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Σε 28. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται τροπολογία 1133 της παραγράφου 58α νέας άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 1134 επί της 58α νέας άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 11.35 επί της παραγράφου 58β νέας άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται συμβαστική σε ΙΟ 25 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται σε ΙΟ 26 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας της ψηφοφορία εγκρίνεται. Τροπολογία 1143 της παραγράφου, επί της παραγράφου 61 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 1149 επί της παραγράφου 62 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 1151 επί της παραγράφου 63 άρχεται η ψηφοφορία. πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 1150. Επί της παραγράφου 63 πάντοτε άρχεται η ψηφοφορία. Πέραση ψηφοφορίας απορρίπτεται. Ε, επί της παραγράφου 3α 1152 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 1153 επί της παραγράφου 63α νέας άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 1154 Επί της παραγράφου 63β νέας ναι, άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβαστική σε ΙΟ 27 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 1163 της παραγράφου 65 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. Υπάρχει μια προφορική τροπολογία της Μόνικα. Ωραία. Τη γνωρίζουμε. Άρχεται η ψηφοφορία. <clears throat> Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 11.65 τώρα επί της παραγράφου 65α νέας. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 1166. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 1168 το πάντοτε επί της παραγράφου 66 άρχεται ψηφοφορία, πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται 645 επί της παραγράφου 2α άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται 1169 επί της παραγράφου 67 άρχεται ψηφοφορία Πέραση ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 11.71. Επί της παραγράφου αλφά άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 11.74 επί της παραγραφου τα 67β άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. 11.75 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 1176. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. 1178. Άρχεται η ψηφοφορία για τις παραγράφους 8α. Πέρας. Εγκρίνεται. 1177. Επίσης, της παραγράφου 68 άρχεται η ψηφοφορία, πέρας. Όχι, απορρίπτεται λέει πρόεδρος, απορρίπτεται. Λοιπόν, ε, συμβαστική σε 29 ε άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 11.80, επί της παραγράφου 69 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας Εγκρίνεται. Συμβασική σε ΙΟΕ 30. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται. 11.82. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Συγγνώμη, λέει η πρόεδρος, δεν ήταν το 82, ήταν 1183. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 1184. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 1185. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας Απορρίπτεται. 1187. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. 1200. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία απορρίπτεται. Περάμε στα εξωτερικά σύνορα. Ε, ε, 73, τροπολογία 1201. Άρχεται ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορία, εγκρίνεται. 1202 για την παράγραφο 73 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Η συμβαστική ΕΒ1 άρχεται ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 1205 για την παράγραφο 73 η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται. 1206 παράγραφα 73 σε άρχεται ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική ψηλών Β2. Άρχεται ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται. Τροπολογία 1213 επί της παραγράφου 75 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 1211 επί της παραγράφου 75 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας απορρίπτεται. 1212 επί της παραγράφου 75 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται παράγραφος 75 1214 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται επί της παραγράφου 75α ε, τροπολογία υπαριθμών 1215 άρχεται η ψηφοφορία Πέρας. Απορρίπτεται. Δύο ταυτόσημες, ε, η 1206 και η 1217 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτονται. 1218. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 1219 μέχρι 1222 και πάμε στην ε, παράγραφο 7. Πέρας ψηφορής απορρίπτεται. Ε, Le vote est clos rejeté. 693 απορρίπτεται. Το 730, 736 παράγραφος 10C πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Παράγραφος 77 δύο ταυτόσιμες τροπολογίες 1223-1224 άρχιτε ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. Το 1225 άρχεται η ψηφοφορία, πέρας της ψηφοφορίας, απορρίπτεται. Ε, συμβαστική ΕΒ4, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 12.33, 12.34, 12.35 και 12.36 και 12.37 ταυτόσιμες. Επί της παραγράφου 79 άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. 1249, επί της παραγράφου 80, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίες, απορρίπτεται. Η 1249, 1240, 1241, επί της παραγράφου 80, είναι ταυτόσιμες, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίες, απορρίπτεται. 1242, άρχεται η ψηφοφορία Πέρας της ψηφοφορίας απορρίπτεται. 1243 και 1244 ταυτόσιμες. Άρχεται ψηφοφορία επί της παραγράφου 81. Πέρας ψηφοφορίας απορρίπτεται. Η 1246 Άρχεται ψηφοφορία για την 81. Πέρας ψηφοφορία, απορρίπτεται. 1245 Άρχεται ψυχοφορία, ψηφοφορία. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 1247 επί της παραγράφου 82 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψυχοφορίας, ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. 1248. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας ψυχοφορίας απορρίπτεται. Συμβαστική ΕΒ5 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβιβαστική ΕΒ6 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. 1254 ταυτόσιμη με την 1255 και 1256 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται η 1257 α όχι καταπίπτει λέει πρόεδρος 1258 από τις παραγράφου 85α άρχεται η ψηφοφορία πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται η 1259 άρχεται η ψηφοφορία πέρα τη ψηφοφορία. απορριπτεται Απορρίπτεται. Συμβαστική ε7 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορια εγκρινεται εγκρίνεται. Συμβαστική ε8 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορια εγκρινεται εγκρίνεται. Συμβαστική ε9 άρχεται. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. ΕΒ10 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβαστική ήταν ΕΒ11 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική ΣΕΤΕ F1. Ψηφίζουμε. Πέρας. Εγκρίνεται. CTF2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1303 της 92. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Τέλος. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1305, παράγραφος 93, άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. Τροπολογία 1307 και 1308 για την παράγραφο 94. Τι, τι συνέβη? Ίσως να αλλάξετε θέση, μήπως. Ωραία. Τροπολογία 1307-1308, ταυτόσημε σε επί της παραγράφου 94. Ψηφίζουμε. Πέρας. Απορρίπτονται. 1309. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 1310. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Πάντα επί της παραγράφου 94. Πέρας ψηφοφορίας. Απορρίπτεται. Συμβιβαστική CTF3. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται CTF4. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Τέλος εγκρίνεται Τροπολογία 1316 επί της παραγράφου 96α. Ξεκινάμε. Τέλος. Εγκρίνεται. 1318 για την παράγραφο 96c. Ξεκινάμε. Τέλος. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική CTF5. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 1324. Παράγραφος 97. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Τέλος. Η ισοψηφία άρα απορρίπτεται. Μα τι συμβαίνει. 1326 ξεκινάει η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνατε. CTF 6 ξεκινάει η ψηφοφορία. Τέλος αυτής εγκρίνεται. CTF 7 ξεκινάμε. Τέλος εγκρίνεται. CTF 8 ξεκινάμε. Τέλος εγκρίνεται. CTF 9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1340 γιατί την παράγραφο 99α. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 1345 για την 99α. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Τέλος. Εγκρίνεται. 1347 παράγραφος 99β. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε τώρα στο συμβαστικό πακέτο για τις δημόσιες υποδομές. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρας αυτής. Εγκρίνεται. Άρα, μέσω αυτής της ομαδικής εγκρίσεως, μπορούμε να πάμε πού να πάμε. Στο πακέτο για τους πρόδρομους ουσίες εκρηκτικά, πρόδρομους εκρηκτικών. Εντάξει, φτάσατε εκεί. Το βρήκατε. Ξεκινάει η ψηφοφορία για τη συμβαστική, για τις πρόδρομες ουσίες, για τα εκρηκτικά. Άρχεται. Πέρας ψηφοφορίας εγκρίνεται και προχωράμε και πάμε στη δέσμη περί παρανόμου εμπορίων, εμπορίου πυροβόλων όπλων. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας αυτής. Εγκρίνεται. Πάμε στην τροπολογία 1406. Επί της παραγράφου 121α. Εντάξει, ψηφίζουμε. Τέλος. Εγκρίνεται. 1411. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Πάμε στην 1420. D. Για την παράγραφο 123. Άρχεται. Πέρας. Απορρίπτεται. 1421. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. 1422. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 1423. Α, καταπίπτει. Συγγνώμη, συγγνώμη, λέει Πρόεδρος. Πάμε στην 1424. Α, έγινε λάθος. Να επαναλάβουμε, αν δεν υπάρχει αντίρρηση. Δεν υπάρχει αντίρρηση να ξανακάνουμε λοιπόν την 1422. Ξαναψηφίζουμε την 1422 για την παράγραφο 123. Ξεκινάμε. 1422. Πέρας. Απορρίπτεται μέσω ε, ισοψηφίας. 1423 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. 1424 και 1425 και 1426 είναι ταυτόσιμες. Ψηφίζουμε για την παράγραφο 124. Πέρας. Απορρίπτονται. 1427. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. 1428 άρχεται η ψηφοφορία. 1428 άρχεται η ψηφοφορία. Ψηφίστε παρακαλώ. Τέλος. Απορρίπτεται. Συμβαστική ED1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1433. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 1434. Για την παράγραφο 125α. Ξεκινάει η ψηφοφορία. 1434. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Τέλος ψηφοφορίας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική ED2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 1437, παράγραφος 125, Β. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας αυτής. Απορρίπτεται 1438 για την παράγραφο 125 Β. Άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 1442 επί παραγράφου 125D άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 1444 άρχεται η ψηφοφορία πέρας ισοψηφία απορρίπτεται παράγραφος των θυμάτων. Συμβαστική V1. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική V2. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. V3. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1463, για την παράγραφο 128α. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 1464. Άρχεται η ψηφοφορία για την παράγραφο 128α. Πέρας. Εγκρίνεται. 1465. Ξεκινάει η ψηφοφορία μας. Τέλος. Εγκρίνεται. 1466 ξεκινάει η ψηφοφορία επί της παραγράφου 129. Πέρας. Εγκρίνεται. 1467 άρχεται η ψηφοφορία επί της παραγράφου 129α. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική Β4 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 1471 επί της παραγράφου 131 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας αυτής εγκρίνεται. Συμβιβαστική V5 άρχεται η ψηφοφορία. Τέλος εγκρίνεται. 1475 επί της παραγράφου 133 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 1476 επί της παραγράφου 133 α άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 1477. άρχια της ψηφοφορία. Επί της παραγράφου 133α. Πέρας. Εγκρίνεται. 1478. άρχια της ψηφοφορία. Επί της παραγράφου 133β. Πέρας. Εγκρίνεται. 1479. Επί της παραγράφου 133c. Πέρας εγκρίνεται. 1480, επίσης παραγράφου 134, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας αυτής απορρίπτεται. 1482 ξεκινάει η ψηφοφορία για την παράγραφο 134. Πέρας εγκρίνεται. 1486 ξεκινάει η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. 1485 ξεκινάει η ψηφοφορία. Τέλος. Απορρίπτεται. 1487 άρχεται η ψηφοφορία πέρας απορρίπτεται 1484 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 1440 άρχεται η ψηφοφορία πέρας εγκρίνεται 928 Άρχεται η ψηφοφορία για την παράγραφο 28α. Πέρας. Απορρίπτεται. 1489 επί της παραγράφου 135α άρχεται. Πέρας. Α, περας απορριπτεται 1489 επι της παραγραφου 135 α αρχεται περας απορριπτεται 1488 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. 1492 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απορρίπτεται. Πάμε στα θεμελιου δικαιωματα δικαιώματα. Συμβαστική FR6. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Περνάμε στη FR5, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 1491, τροπολογία 1491 επί της παραγράφου 136, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 619, άρχεται η ψηφοφορία. Απερίφθη. Τροπολογία 1504 επί της, επί της παραγράφου 136α άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται και περνάμε στη 1507. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Εφέρ FR7. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρας εγκρίνεται συμβιβαστική FR8 άρχεται πέρας εγκρίνεται τροπολογία 1511 άρχεται η ψηφοφορία αφορά την ε, παράγραφο 137α απερίφθη και περνάμε στη συμβαστική FR9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 1514 επί της παραγράφου 138α. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Συμβιβαστική FR10. Συγγνώμη, 10 αρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Τροπολογία 621, παράγραφος 1C, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας, απερίφθη. Τροπολογία 1144, διονομαστικής κλίσεως, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας, απερίφθη. Συμβιβαστική ΕΦΕΡ 11. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 15-18. Άρχεται η ψηφοφορία. Μην τρώτε μόνο σας, λέει η Πρόεδρος, δώστε και σε μας. Άρχεται η ψηφοφορία τώρα. Πέρας της ψηφοφορίας. Απερίφθη. 15-19, παράγραφος 139α, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Αιτιολογικές αναφορές, 1, τροπολογία 1, άρχεται η ψηφοφορία. Απερίφθη. Τέσσερα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Περνάμε τώρα στην συμβιβαστική IF5. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβιβαστική IF6 άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Ε, δεν θα διακόψουμε, λέει η Πρόεδρο. Συνεχίζουμε. Ε, IF7 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα της ψηφοφορίας εγκρίνεται. IF 8. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 35. Αιτιολογική σκέψη D. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Συμβιβαστική IF 9 Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική IF10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική IF11. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Ε, τροπολογία 55. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβαστική IF 12. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 62. 62. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία, αλλά απερίφθη. Τροπολογία, συγγνώμη, 63. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Συμβιβαστική IF 13. Άρχεται η ψηφοφορία. πέρας. Εγκρίνεται τροπολογία 70, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Συμβιβαστική T6 για την τρομοκρατική απειλή. Ψηφίζουμε. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Συμβιβαστική T7 άρχεται η ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τροπολογία 89 άρχεται. Πέρας απερίφθη. Συμβιβαστική T8 άρχεται. Πέρας Εγκρίνεται. Τροπολογία 96. Άρχεται η ψηφοφορία. Απερίφθη η τροπολογία. Τροπολογία 116. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Συμβαστική T9. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας εγκρίνεται. Συμβαστική T10. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Και πάμε στην T11. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία υπεριθμών 125. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία συμβιβαστική Т12. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Περνάμε στη συμβαστική T13. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Και εγκρίνεται. Τροπολογία υπαριθμών 140. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 141. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 143. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 144. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας και απερίφθη. 145. Άρχεται. Πέρας. Απερίφθη. 146. Άρχεται η ψηφοφορία. Εκατόν 147, 148 ταυτόσημες. Ψηφίζουμε λοιπόν. Απερίφθη. Τροπολογία 150 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 149. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται. Τροπολογία 151. Α, όχι. Περνάμε στη συμβαστική T15. Άρχεται. Το 151 είχε καταπέσει και ψηφίζουμε την συμβαστική T15. Πέρας της ψηφοφορίας εγκρίνεται. Τροπολογία 160 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Απερίφθη. Τροπολογία 161. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. Συμβιβαστική T16. Άρχεται. Πέρας εγκρίνεται. Τροπολογία 167. Άρχεται η ψηφοφορία αφορά την αιτιολογική σκέψη TA. πέρας της ψηφοφορίας, απερίφθη μάλιστα. Τροπολογία 168. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Εγκρίνεται. 169. Άρχεται. Πέρας. Εγκρίνεται συμβιβασμοί